Τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης θα υποβληθούν στην προσεχή συνεδρίαση προς έγκριση. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, λύεται η συνεδρίαση. Διακόπτονται οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συνεδρία Ολομέλειας, λύεται η συνεδρίαση.